Σας ευχαριστώ. Τα πρακτικά της θεσινής συνεδριάσεως είναι στη διαθεσή σας. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με την έκθεση της κυρίας Ματέρα